πλέον και το δήλωσε στην αντίστοιχη αντιπροσωπεία. Προχωράμε τώρα με τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα συμπεράσματα τη διάσκεψη των ΕΕ για το ρατσισμό Ντέρμαν 2. Κύριε ε, εκπρόσωπε του Συμβουλίου, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για την ευκαιρία που μας δίνετε για να αναφερθώ στη διάσκεψη του ΟΗΕ που γνωρίζω ότι παρακολουθούν πολλοί βουλευτές από στενά. Η προκαταρκτική διαδικασία της διάσκεψης ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκη με πολλές χώρες να έχουν σοβαρές αμφιβολίες για την διαδικασία ειδικά μετά τα γεγονότα του 2001 λόγω των ανησυχιών για το ότι θα εκφραστεί θα χρησιμοποιηθεί η διάσκεψη για την έκφραση απόψεων μη ανεκτικότητα πολλα πολλά κράτη-μέλη όπως και το δικό μου αποφάσισαν να μην παραστούν. Πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε από την παρέμβαση ενός μέλους στην αρχή της διάσκεψης. όχι μόνο ήταν εντελώς απαράδεκτο, αλλά ήταν και τελείω αντίθετο με το πνεύμα της διάσκεψης. Είναι ατυχές αν και ίσως αναπόφευκτο, πως το γεγονός αυτό και η αποχώρηση όλων των κρατών μελών της Ένωσης και άλλων μελών του ΟΗΕ εμπόδισε την συνενετική οθέτηση του τελικού εγγράφου. Ταυτόχρονα θεωρώ πως η πολύ επικοδομητική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προπαρασκευαστική φάση της διάσκεψης πρέπει να αναγνωριστεί. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά τη σύνταξη του τελικού εγγράφου στο οποίο έπαιξε κρίσιμο ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά τα γεγονότα στα οποία αναφέρθηκα, το γεγονός πως το τελικό έγγραφο της διάσκεψης σέβεται όλες τις κόκκινες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί σοβαρό επίτευγμα. Το τελικό έγγραφο σέβεται πλήρως το υπαρκτό πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης και συμμορφώνεται με πολλά από τα αιτήματά μας όπως την ανάγκη να αποφευχθεί οποιαδήποτε αναφορά στην ε, δυσφήμιση θρησκειών και συγκεκριμένα μεμονωμένη καταδίκη του Ισραήλ. Ειδικά παρέμεινε η παράγραφος καταδίκης του ολοκαυτώματος. Πρέπει τώρα να σκεφτούμε ποια είναι τα αποτελέσματα και για την Ένωση και για το τελικό έγγραφο. Θα συνεδριάσουμε ιδιαίτερα για να ορίσουμε το πώς θα εφαρμόσουμε τις δεσμεύσεις οι οποίες έχουν αναλυφθεί. Το Συμβούλιο ανισχύει ιδιαίτερα από τα φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας τα οποία θεωρούμε τι σοβαρότερε προκλήσεις σήμερα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γνωρίζω πως συμφωνεί μαζί μας το Κοινοβούλιο και έχετε παίξει κέριο ρόλο στο να δημιουργήσετε την νομοθετική βάση και τα πρακτικά εργαλεία για να καταπολεμηθεί αυτή η μάστιγα. Η καταπολέμηση του ρατσισμού είναι μια πρόκληση που απαιτεί συνεχή πρακτικά μέτρα και στον τομέα της εκπαίδευσης. Επίσης, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης και να προωθηθεί η ανεκτικότητα. Ενώ υπάρχουν σημάδια πως σχετική νομοθεσία της Ένωσης έχει θετικό αντίκτυπο, η γενική παγκόσμια πρόοδος δυστυχώς παραμένει αργή υπάρχει μια τάση σε πολλές χώρες που είναι μάλιστα αρνητική. Έχουμε δει περιπτώσεις στις οποίες η οικονομική κρίση προκαλεί ρατσιστικές ε, τάσεις και τάσεις ξενοφοβίας. Οπότε απαιτούνται τώρα ισχυρότερες αντιρατσιστικές πολιτικές και εντός της Ευρώπης και ευρύτερα αντιμετωπίζουμε αύξηση της βίας κατά προσφύγων και τον τον άσυλο καθώς και μειονοτήτων όπως η Ρώμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ισχυρό και εκτιμένο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και τα δύο αυτά φαινόμενα είναι ασύμβατα με τις αρχές ε, στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταδικάσει επανειλημμένα κάθε μορφή ρατσισμού και θα συνεχίσει να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των εξουσιών που έχει από τις συνθήκες θα συνεχίσει να καταπολεμά το ρατσισμό και την ξενοφοβία και εντός της Ένωσης και στο πλαίσιο της εξωτερικής μας δράσης. Εσωτερικά έχουμε υιοθετήσει νομοθεσία που απαγορεύει την άμεση και έμεση διάκριση με βάση την φυλή ή την εθνοτική καταγωγή στην εργασία και την εκπαίδευση και την πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες. Επίσης απαγορεύεται η διάκριση για άλλους λόγους μεταξύ των οποίων η θρησκεία, η ηλικία, σεξουαλικός προσανατολισμός και αναπηρίες, ειδικά στην εργασία. Επίσης έχουμε υιοθετήσει νομοθεσία που απαγορεύει τα κηρύγματα μίσους και την παρακίνηση σε βίαιες πράξεις κατά μιας ομάδας, ειδικά όταν η ομάδα αυτή ορίζεται από τον φιλή γλώσσα και τα λοιπά. Ναι. Επίσης δεν επιτρέπεται το να μειώνει κανείς την έκταση των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Τα ζητήματα αυτά λοιπόν στον διμερή πολιτικό διάλογο με τις τρίτες χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα επίσης προωθούνται και διασφαλίσαμε πως ο ρατσισμός και η ξενοφοβία ενσωματώνονται στις στρατηγικές μας της συνεργασίας όπως η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας πολλά συμβαίνουν σε πολυμερή φόρα, π.χ. στον ΟΑΣΕ. Συντονιζόμαστε τα κράτη-μέλη για να διασφαλίσουμε πως ε, οι δεσμεύσεις των 56 κρατών μελών του ΟΑΣΕ γίνονται σεβαστές. Το ίδιο συμβαίνει και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στο ευρύτερο πλαίσιο του ΟΗΕ. Τα παραδείγματα αυτά καταδεικνύουν την συλλογική μας δέσμευση για να εργαστούμε σε αυτό το ζήτημα και εσωτερικά και εξωτερικά. Η διάσκεψη του Ντέρμπαν ήταν μέρος αυτής της διαδικασίας, δεν ήταν εύκολο και σαφώς σημαδεύτηκε από αυτούς που θεώρησαν ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν τη διάσκεψη για τους δικούς τους σκοπούς, αλλά στο τέλος επικεντρώθηκε η προσοχή μας και στην ανάγκη να αντιμετωπίσουμε το ρατσισμό και την ε, ξενοφοβία και στην δέσμευση την οποία έχουμε αναλάβει και εμείς και πολλοί άλλοι για να εξαλειφθεί αυτή η μάστιγα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Ζακμπαρό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτέ. Χαίρομαι που μου δίδεται η ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτή την συζήτηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολούθησε από πολύ κοντά τα, τις προετοιμασίες και την προπαρασκευή της διασκέψεως του Ντέρμπαν έτσι ώστε να προετοιμαστεί σωστά η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη διάσκεψη. Λάβαμε υπόψη μας κατά αυτή την έννοια την ε, έκκληση ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δέσμευε, που καλούσε την Ευρωπαϊκή, την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει ενεργά στην εξέταση της σκέψης του ε, Ντέρμπαν. Η, όσον αφορά τα συμπεράσματα και όσον αφορά ε, την συνέχιση του ψηφίσματος που είχατε εγκρίνει την 19η Ιανουαρίου. Όπως ξέρετε, πέντε κράτη-μέλη αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στη διάσκεψη αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ε, παρόλα αυτά να παραμείνει ως παρατηρήτρια γιατί συμμερίζεται την άποψη της πλειοψηφία των κρατών μελών, σύμφωνα με τις οποίες οι κόκκινες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελικά διατηρήθησαν στο κείμενο της διάσκεψης. Στο τελικό κείμενο, το οποίο αποτέλεσε απόρρια ενός συμβιβασμού και κατά αυτή την έννοια δεν μπορεί να είναι ένα ιδεώδε κείμενο, παρόλα αυτά το έγγραφο αυτό δεν περιέχει κανένα στοιχείο συκοφάντηση είτε αντισημιτικού χαρακτήρα, είτε οποιαδήποτε συκοφάντηση χωρών σε οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου, είτε οποιαδήποτε συκοφάντηση ε, θρησκειών. Η τελική έγκριση του εγγράφου από 182 χώρες ε, μέλη των Ηνωμένων Εθνών επιβεβαιώνει την βούληση της ε, ε, κοινής, την, βούληση των κρατών σε όλο τον κόσμο να πολεμήσουν ενάντια στον ρατσισμό και βεβαίως απεφεύχθη η προσπάθεια εγχειρηματοποίησης της διασκέψεως για λόγους αντισημιτικούς. Εν πάση περιπτώσει, τα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα στη διάρκεια της ε, διάσκεψης δεν ε, μειώνουν με κανένα τρόπο τις προσπάθειες που έχει μέχρι τώρα καταβάλει και θα εξακολουθήσει να καταβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να καταπολεμήσει οποιαδήποτε μορφή και οποιοδήποτε είδους ξενοφοβία και ρατσισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τον αγώνα της καλά, κατά της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και του αντισημιτισμού εντός και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και βεβαίως ε, στο μέτρο των ε, ε, δυνατοτήτων που τις παρέχονται από τις συνθήκες. Και πρέπει να σας πω κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ, ότι προσωπικά εγώ θα παρακολουθήσω προσεκτικά και στενά την υλοποίηση της απόφασης πλαίσιο ρατσισμός και ξενοφοβία από τα κράτη-μέλη. Δεσμεύομαι προσωπικά σε αυτήν την εποπτεία και την παρακολούθηση όσον αφορά ε, την ενσωμάτωση αυτής της ε, απόφασης πλαισίου και οφείλω να ομολογήσω ότι η υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι ένα μέσο που έχουμε και εμείς πλέον στη διάθεσή μας έτσι ώστε να παρατηρούμε και να παρακολουθούμε με σταθερότητα τα φαινόμενα αυτά. Είναι γεγονός βεβαίως ότι μπορούμε να ευχηθούμε μελλοντική διάσκεψη ε, των Ηνωμένων Εθνών για το ρατσισμό να μην στιγματιστούν από αυτή αυτά ε, τα απαράδεκτα στοιχεία και από αυτήν την παρένεση προς την βία και τον ρατσισμό, αλλά σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι το αποτέλεσμα ήταν αρκετά ικανοποιητικό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντεπρόεδρε. Ξεκινάμε με τους αγορητές εξ ονόματος των ομάδων. Από πλευράς ΕΛΚ ο κύριος Τάνοκ. Ο Ιρανό πρόεδρο Αχμαντινιτζάν πρόσφατα στη διάσκεψη του ΟΗΕ στη Γενέβη για τον ε, κατά του ρατσισμού είπε ότι το Ισραήλ ε, ε, είναι ρατσιστική χώρα. Δημαγωγικά μίλησε τραβώντας τα φώτα της δημοσιότητας πάνω και ζήτησε βέβαια και το σβήσιμο από το χάρτη της χώρας αυτής και ότι έχει πυρηνικά όπλα, κάτι το οποίο επιθυμεί και η ίδια όμως η χώρα του να αποκτήσει. Πολύ σωστό όμως κατά την άποψή μου το Ισραηλινό κράτος αποτελεί εταίρο και σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, στόχος ε, ε, είναι να δούμε υπάρχει άλλη χώρα πολιτισμικότερη και με έκφραση όλων των θρησκειών από το Ισραήλ. Σίγουρα το Ισραήλ διατηρεί μια ανοιχτή μεταναστευτική πολιτική είναι ε, το σπίτι όλων των ε, Εβραίων ανά τον κόσμο αλλά και η αραβική κοινότητα απολαμβάνει των δημοκρατικών ε, δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. ποπτέύουμε ότι ο Αχματινετζάν αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να μεταστρέψει την προσοχή από το αποτροπιαστικό ιστορικό καταπατήσεων των Ευρωπαϊκών δικαιωμάτων στη χώρα του που δεν υπάρχει ελευθερία των δημοσιογράφων ότι ο ίδιος μιλά για την ελευθεροτυπία, ακόμη και φρικτές εκτελέσεις και διαλυθοβολισμού. Οι μειονότητες ε, όπως οι χριστιανοί παραδείγματος χάρη που διώκονται, ενώ στο Ισραήλ ε, οι μειονότητες γίνονται σεβαστές και τα δικαιώματά τους σε σεβαστά επίσης. Δεν θα πρέπει λοιπόν ε, να κατηγορούμε το δημοκρατικό εταίρο μας, το Ισραήλ, αλλά τις βαρβαρότητες του Ιρανικού καθεστώτος. Εγώ είμαι υπέρ ε, της ε, μετριοπάθειας και κατά του φανατισμού. Είναι καλό να φροντίσουμε στο μέλλον ο Αχμαντινετζάν να αποέχει από τέτοιου είδους συνεδριάσεις και να μην λέει αυτά που λέει. Εκ μέρου τη Σοσιαλιστική ομάδα τώρα η κυρία Γκόμε για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να θεωρήσουμε επιτυχές ε, το συνέδριο στο Ντέρμπαν. Έχουμε τις πέντε κόκκινες γραμμές ε, που όρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο έγγραφο αυτό και επίσης αντικατοτρίζεται σε αυτό μία σαφής ε, συνένεση. Δυστυχώς όμως το έγγραφο αυτό δεν θα μείνει αυτό χαραγμένο στη μνήμη όσων ε, παρέστησαν ε, στις συζητήσεις της Γενέβης. Υπήρξαν βαθιοί διχασμοί ε, για ένα συνέδριο το οποίο ήταν αφιερωμένο σε ένα θέμα όπως η καταπολέμηση του ρατσισμού. Η Ευρώπη για μια ακόμη φορά έδειξε πόσο εύθραυστη είναι και η ενότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά ακόμη μπορεί απέχει από το να είναι συμπαγής όσο θα θέλαμε. Το σημαντικότερο νομίζω θα ήταν όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση να βγει συλλογικά εκτός αίθουσας ακούγοντας τα προκλητικά και απαράδεκτα λόγια του κυρίου Αχμαντινετζάντ. ο οποίος ήρθε σε σύγκρουση με τις ε, σημαντικότερες χώρες της Δύσης. Ο μοναδικός στόχος άλλωστε της ομιλίας του ήταν να κατηγορεί, να διαιρεί και να προκαλεί. Όμως η τη ενώση και παρόλα αυτά εμείς δείξαμε αδυναμία, δείξαμε ότι είμαστε διαιρεμένοι ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε απαντήσει πιο καλά στις προκλήσεις του Αχμαντινέτζα. κυρία Ιντβελ τώρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να κάνω μια γενική φύσεως παρατήρηση. Οι χώρες δεν είναι ρατσιστικές, οι άνθρωποι είναι ρατσιστές. Και είμαι βεβαία ότι στο Ιράν υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν συμμερίζονται τις απόψεις του Προέδρου τους. Και επομένως ε, χάσαμε μια καλή ευκαιρία να δείξουμε ότι η Ευρώπη δεν είναι σιωπηλή, ότι η Ευρώπη είναι παρούσα και ότι μπορεί να ορθώσει το αναστημά και να μιλήσει εξ ονόματος αυτών των ανθρώπων που δεν συμφωνούν με τον πρόεδρό τους. Εγώ προσωπικά ήμουν κατά του καθαρίσματος ε, της ε, διάσκεψης. Αλλά βέβαια αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε ευρωπαϊκή στρατηγική. Γιατί ήταν χωρισμένη η Ευρώπη, γιατί άραγε και θα ήθελα να μου πει το Συμβούλιο και μάλιστα εγώ έχω υποβάλει κατά αυτή την έννοια ε, μία τροπολογία στην έκθεση Ραϊμόνο Μπιόλς την οποία θα συζητήσουμε σε λίγο. Γιατί η Ευρώπη ε, των 27 χωρών δεν, μπορούν να δεν μπορεί να συμφωνήσει ε, επί μιας κοινής στρατηγικής. Εάν το Συμβούλιο ε, ε, κοινοποιήσει ένα έγγραφο, επ' αυτού θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι 27 χώρες. Ε, επομένως, δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να συμφωνούμε επί μιας κοινής θέσης. Απ' την άλλη πλευρά, όσον αφορά την συκοφάντηση των θρησκειών, ε, μου κάνει εντύπωση που υπάρχει ένα κείμενο των ΗΠΑ που απαγορεύει την συκοφάντηση των θρησκειών. Ε, βλέπω, διαβλέπω όμως και την ηρωνία, δηλαδή ότι εδώ στο σώμα μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ασκήσει κανείς κριτική. Προσέξτε, όχι να μιλήσει κατά ή να καταδικάσει, να, να, να επικρίνει, να, δείξει η επικριτική στάση απέναντι σε κάποια ε, θρησκεία. Ε, και βεβαίως ε, εγώ μαζί με άλλους συναδέλφους μου έχω καταδικάσει ήδη την τοποθέτηση του Πάπα όσον αφορά την χρήση προφυλακτικών που σαφώς αντιτίθεται στον αγώνα για την καταπολέμηση του AIDS. Πρόεδρος, θα ήθελα να σας ζητήσω ότι να σας ζητήσω λοιπόν να μην υπερβαίνετε το χρόνο σας γιατί το πινάκιο του συνεδρία συνεδρίασης είναι εξαιρετικά βεβαρημένο. Catch the eye. Τώρα έχω δύο. Αντρίκενε, η κυρία Αντρίκενε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω για μία ακόμα φορά ότι το τελικό κείμενο ε, της διάσκεψης αναθεώρησης του Ντέρβαν ε, έγινε, δεκτό με συνένεση και κατά πλειοψηφία. Έστω και αν δεν είναι το ιδεώδες κείμενο, αποτελεί ε, τη συμβαστική λύση μετά από μία διαπραγμάτευση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση, να συνεχίσουμε και να ανοίξουμε συζήτηση για το νέο, το νέο έγγραφο έτσι ώστε ε, θέματα όπως ο ρατσισμός, ε, η ξενοφοβία, τα κλισέ, τα στερεότυπα ε, και οι προκαταλήψεις να πάψουν. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω συζήτηση με μη πολεμικό χαρακτήρα και ε, πρέπει να πούμε ότι η διαδικασία του Ντέρμπαν ε, θα πρέπει να συνεχιστεί χωρίς ε, ιδεολογίες και ιδεολειψίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, να καταπολεμήσει τον ρατσισμό και την ξενοφοβία και θα πρέπει να δούμε μήπως τελικά η διάσκεψη του Ντέρμπαν πηγαίνει προς τη λάθος κατεύθυνση. Ναι, βεβαίως ε, είναι προφανές και είναι κρίμα που τα ε, θύματα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας ε, δεν είχαν την θέση τους σε αυτήν την διάσκεψη. Έγινε μια προσπάθεια η οποία επιτεύχθη στο τέλος παρέκκλησης ε, τη διάσκεψης ε, του ε, Ντέρμπαν από τον πρόεδρο του Ιράν και πολλοί έπεσαν στην παγίδα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τις χώρε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης που έμειναν και που δεσμεύτηκαν και που τελικά μας έδωσαν την δυνατότητα να ακούσουμε κάποια συμπεράσματα τα οποία μπορεί να μην είναι τα ιδεώδη. Ένα κείμενο μπορεί να μην είναι το ιδεώδε, αλλά τουλάχιστον υπάρχει. Και θα ήθελα να μου πει, ε, να ακούσω διαστόματο της Προεδρίας ε, τι τους οδήγησε αυτή την εκτρή στάση η οποία ε, διαμέλησε στου πέντε ορίζοντες την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εμπλακεί πλήρως και στην προετοιμασία της διάσκεψης και στη σύνταξη του τελικού εγγράφου με στόχο να γίνει όσο δυνατόν πιο ισορροπημένο και να σέβεται τις υπάρχουσες διατάξεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης. Επίσης, επέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αναφερθεί μεμονωμένα το Ισραήλ. Οπότε τελικά καταφέραμε ένα κείμενο που σεβόταν τις δικές μας κόκκινες γραμμές, ανεξαρτήτως του ότι κάποια κρατημέλη αποφάσισαν να μην ε, συμμετάσχουν υπό την, ε, εθνική, την τους ε, ιδιότητα. Αυτό όμως δεν εμπόδισε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκφραστεί ως Ένωση. Η Προεδρία συνέχισε τον εσωτερικό συντονισμό που συμπεριλάμβανε και την ε, προετοιμασία δύο δηλώσεων, μία εξ ονόματος ε, της Σουηδίας. που εκφώνησε και τις δύο Σουηδίας ε, και ε, εκφωνήθηκαν και οι δύο από τη Σουηδία που είναι η επερχόμενη Προεδρία. Βεβαίως η μη συμμετοχή μας θα έθετε να αμφιβόλω την δεσμευσή μα για να αγωνιστούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε ένα στέρεο κεκτημένο στο οποίο θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε όπως σωστά επισημάνθηκε. Δέχομαι την κριτική αυτή. Δεν καταφέραμε τελικά να βρούμε έναν κοινό τόπο. Δεν υπήρχε κοινό τόπο, οπότε δεν υπήρχε και θέση κοινή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αποφασίστηκε να τοποθετηθούν οι χώρες με τις εθνικές τους θέσεις και εκπροσωπήθηκαν ως χώρες μεμονωμένες στα καρτιμένη. Αλλά οφείλω να πω αυτό το οποίο τονίσαμε και στην τελευταία συνεδρίαση. Οι υπουργοί συζήτησαν αυτό το ζήτημα, θα λύσουν τα διδάγματά τους και θα πρέπει να επανέλθουν βεβαίως σε αυτό το θέμα γιατί δεν ήταν και ηρωική ακριβώς η στάση μας στη διάσκεψη αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ όλους ε, όσους πήραν το λόγο. Την ε, προηγούμενη Δευτέρα η Επίτροπος Φεραίρο Βάλνερ ε, συναντήθηκε με τον ύπατο αρμοστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, του, των Ηνωμένων Εθνών στα πλαίσια διάσκεψης σε επίπεδο Υπουργών των Ηνωμένων Εθνών και επανέλαβε αυτά που είχε πει στις 8 Οκτωβρίου 2008 στις Βρυξέλλες σε μία διάσκεψη που είχε συνοργανωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, σχετικά με την προστασία αυτών που ε, ε, ε, υπεραμείνονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εξεφράστη η άποψη ότι θα πρέπει σε όλο τον κόσμο να υπεραμεινθούμε των δικαιωμάτων του ανθρώπου γι' αυτό λοιπόν και η ΥΠΕΤΗ καλεί όλο τον κόσμο να συμμετάσχει σε αυτόν τον αγώνα κατά του ρατσισμού, κυρίως κατά την έννοια του τελικού εγγράφου του Ντέρμπαν. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σκεφτεί πολύ απαντώντας σε αυτήν την πρόσκληση. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επαγρυπνά. Θα πρέπει να είναι προσεκτική έτσι ώστε η στάση της απέναντι σε αυτά τα θέματα να παραμείνει αποτελεσματική. Σημερίζομαι την, ε, ε, τις απόψεις που εξεφράστησαν εδώ από προσωπικής απόψεως ε, και εγώ θεωρώ ότι η Ευρώπη ε, εάν ήταν πραγματικά ενωμένη και δεν είχε διαλυθεί ε, σε επίπεδο κρατών μελών οπωσδήποτε θα μπορούσε να είχε μιλήσει με μία φωνή και επομένως η διαμαρτυρία της απέναντι σε απαράδεκτα λόγια θα ήταν πιο σημαντική αλλά ε, συμφωνώ και υπογραμμίζω αυτά που είπε η Πρόεδρος ότι θα πρέπει αυτό να μας γίνει μάθημα και ελπίζω ότι η θέση μας ενισχυμένη και από, το, από την υπογραφή της συνθήκης της Λισαβόνας θα ενδυναμώσει την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα και επομένως ε, ε, ότι θα είναι και πιο αποτελεσματική και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα και σε διμερές επίπεδο. Ε, και τέλος να ευχαριστήσω τους αγορητές που είπαν πολλά πράγματα με τα οποία συμφωνώ και τελειώνοντας να πω ότι πραγματικά θα πρέπει αυτό το το σημείο να αποτελέσει σημείο ε, σκέψης και τροφή για ε, σκέψη στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν ε, το σημείο αυτό. Τώρα θα συζητήσουμε την έκθεση Ρεμόνο Μπιόλ Σίχερμα, ετήσια έκθεση 2008 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Βλέπω ότι ο κύριος Ομπιόλ φτάνει την κατάλληλη στιγμή, γι' αυτό λοιπόν του δίνω και το λόγο. Κύριε Ομπιόλ, έχετε το λόγο, είστε εισηγητής για